Ευχαριστούμε τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Ξεκινούμε τις ψηφοφορίες. Θα είναι μακροσκελής η ψηφοφορίες, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξεκινάμε με την έκθεση Γκάγερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Απόφαση περιπτώνα. Περιμένουμε να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Να δούμε την πρόταση ψηφίσματο. Τροπολογία 1 υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχέ. απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 άρχεται την ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται, μου φαίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για την 24 ψηφίζουμε, έρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Μάλλον όχι για την 38. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε. Εάν δεν ε, σηκώνετε τα χέρια, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίφθηκε. 37 υπέρ, κατά, με συγχωρείτε. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντε. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. πέρασε. Απορρίπτεται. 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν απαντήσω. Πέρασε. Απορρίπτεται. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. να άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, να απαντήσω. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, να απαντήσω. Πέρας. Απορρίπτεται. 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν απαντέ, Πέρας. Απορρίπτεται. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποθέσει. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία μου. Εψήφισαν άπαντε πέρα. Απορρίπτεται. 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Τα ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνατε. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Παρακαλώ. Ζητά κάποιο το λόγο. Όχι. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παρακαλώ, κυρία Γιάλα. Ah, Κύριε Πρόεδρε, στο ισπανικό κείμενο εμφανίζεται το Eurojust αντί για Eurostat. Θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα. Θα γίνει αλλαγή. Ευχαριστούμε για τη διευκρινήση. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματο. όπως προέκυψε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Σέμετα, θέλει να πάρει το λόγο. Uh, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Επιτροπή ορίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χορηγήσει απαλλαγή στην Επιτροπή για την εφαρμογή του προπολογισμού του 2011. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Γενικό Εισηγητή Γιάνν Σκάια και στους συντονιστές και σκιώδες εισηγητές των πολιτικών ομάδων με τους οποίους είχαμε επικοδομητική συνεργασία καθ' όλη τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Η ψηφοφορία σας σήμερα αναγνωρίζει ότι συνολικά ο προπολογισμό έχει ε, αντιμετωπιστεί και εκτελεστεί σωστά. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι συμμετέχουν ε, στην χορήγηση και τον έλεγχο των ε, κοινοτικών πόρων πρέπει επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους ούτως ώστε να αξιοποιούνται σωστά οι πιστώσεις. Καλό τους συνομοθέτες να λάβουν όπως πρέπει υπόψη το ψήφισμα επί της απαλλαγής που εγκρίθηκε στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να έχουμε νέο νομικό πλαίσιο χωρίς ε, την απλοποίηση που τόσο χρειαζόμαστε και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να χορηγείται περισσότερη αξία στην ε, χρήση των πιστώσεων. Ευχαριστούμε κύριε Πέτροπη. Προχωρούμε. Κοιτάζουμε την έκθεση Γκάγερ για την ε, απαλλαγή του ελεγκτικού συνεδρίου. 2-13 κατά Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.17 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύνολο ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Γκάγερ. Έκθεση Ορτής Βιλέλα. Απαλλαγή 2011 για το Ευρωκοινοβούλιο. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 10 έχει αποσυρθεί. Πρώτη παράγραφος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Με ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε για την πέμπτη τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έντεκα Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 12 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 8 άρχεται η ψηφοφορία. να άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. 6. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. πέρα Εγκρίνεται. 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Δεν ψηφίζουμε την ένατη τροπολογία. Έγινε ένα λάθος από τη γραμματεία. Πρόταση ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία. Άρχια την ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Παρακαλώ. Κύριε Στάς. Το μικρόφωνο σας. Πρόεδρε, νομίζω, Πρόεδρε, νομίζω ότι η τροπολογία 9 δεν υπευλήθη στην Ολομέλεια. Οπότε θα έπρεπε να ψηφιστεί από την Ολομέλεια. Στον ε, κατάλογο ψηφοφοριών μου λέγεται ότι πρέπει να ψηφιστεί. Λέτε λοιπόν να ψηφίσουμε την ένωτη τροπολογία όχι με ονομαστική ψηφοφορία, έγινε λάθο από τι υπηρεσίε. Με συγχωρείτε λοιπόν. Διανάταση τη κυρώσει υπέρ τη ένωτη τροπολογία. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Έκθεση Σόνταγκαρντ. Απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Ψηφίζουμε για την απόφαση. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται πρόταση ψηφίσματος τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται 6 άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν άπαντες πέρας εγκρίνεται 49 πρώτο τμήμα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Συνολική ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, εποχέ. εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Σόλτεγκαρντ. Και τώρα διακόπτουμε τις ψηφοφορία για την επίσημη σύνοδο. δουλεύω μια